Bonjour à toutes et à tous. Buenos días. Καλημέρα. Σε αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά, ο Πρόεδρος. Dear colleagues, if you may take your... Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε. Welcome to the Libre Committee. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Ιστορικών Υποθέσεων. Πρώτη τακτική συνεδρίαση μετά τη συνεδρία συγκρότησε σώμα. Ξεκινούμε πλέον με τις εργασίες μας. Αλλά σας παρακαλώ να κάνετε λίγη ησυχία. Σήμερα και αύριο έχουμε βαρύ πρόγραμμα. Σήμερα συνεδριάζουμε πρωί και μεσημέρι. Παρουσία δύο επιτρόπων, πολύ σημαντικέ παρουσίες. Ο αρμόδιος για θέματα ασφαλείας King και η αρμόδια νομικά ζητήματα Γιούροβα θα είναι εδώ. Να κάθεστε ησύχω, παρακαλώ, επαναλαμβάνει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ λοιπόν να σημειώσετε το χρονοδιάγραμμα. Ξεκινάμε σήμερα 9 και 4, 11.30 λίγη τακτική συνδρίαση και αρχίζουν οι συντονιστές, 11.30 ώρα και το μεσημέρι θα ξαναξεκινήσουμε στις 3. μέχρι τις 4 και 30. Και αύριο πρωί ξεκινούμε στις 9. μέχρι το μεσημέρι στις 12. Ας εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, καταρχάς. Υπάρχουν αντιρρήσεις, όχι. Σε ό,τι αφορά την ημερήσια διάταξη. Okay. Then... Εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Προχωρώ στις ανακοινώσεις του Προέδρου. Καταρχάς, τα γλωσσικά. Να ζητήσω συγγνώμη για το ότι δεν υπάρχει στα Ιρλανδικά και στα λετονικά σήμερα διερμηνία. Βλέπετε οι υπόλοιποι της γλώσσας σας. Εν συνεχεία έχουμε τις συστάσεις των συντονιστών τις πρέπει να εγκρίνουμε. Σε σχέση καταρχάς με τον κανόνα 205, το άρθρο 205 του κανονισμού. Βλέπετε το σημείωμα για τη συνέντευξη 11η Ιουλίου στα έγγραφά σα. Έπειτα έχουμε τον ορισμό των εισηγητών. Ο υποφαινόμενο καταρχά ω πρόεδρο. Θα αναλάβω την έκθεση για την ε, τελεστική απόφαση του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή, αυτό με την ανταλλαγή δεδομένων ε, για τα στοιχεία καταχώρησης οχημάτων στην Ιρλανδία. Έπειτα έχουμε την Ρομπέρτα Μέτσολα από το ΕΛΚ, η οποία θα είναι εισηγήτρια για τον κανονισμό που αφορά πλαστά και γνήσια έγγραφα online. Πρόκειται για το σύστημα FADO. Μετά έχουμε την κυρία Λις Κούνκη από τους Πρασίνους, η οποία θα είναι εισηγήτρια για το πρόγραμμα δικαιωμάτων και αξιών. Σχετίζεται και με το πολιτισμικό πλαίσιο. Μάγκιντ Μάγκιντ τους πρασίνους. Εισηγητής για την οριζόντια οδηγία περισσότερης μεταχείρισης. Και Κλέρ Ντέιλι, Γκούε. Η τέταρτη ανταλλαγή απόψη είναι το Και τέλος, για τις ε, συντάξεις, ε, ε, για τις γνωμοδοτήσεις, συντάκτες έχουμε καταρχάς την Κουέντολ Ντέλμπο Σκόρφιλ, τους Πρασίνους, θα συντάξει γνωμοδότηση για, την, ε, για το σχέδιο προπολογισμού του 2020. Συμφωνείτε με τους ορισμούς αυτούς. Αν ναι, θεωρούμε ότι εγκρίνονται και προχωρούμε. Στο πρώτο σημείο της μέσιας διάταξης, ε, επί της ουσίας που είναι προβλέπεται για τα επόμενα 40 λεπτά μέχρι τις 10. Είναι η συζήτηση από το Γενικό Περιβολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ναι. για το οικονομικό έτος 2020. Θα εξετάσουμε την γνωμοδότηση αφού ακούσουμε την εισηγήτρια, την κυρία Γκουέντολιν Τέλμπο Κόρφιλτ. Και μετά θα μπορούμε να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων ε, μεταξύ των σκιωδών εισηγητών, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όποιο άλλο συναδέλφου θέλει το λόγο. Η εισηγήτρια καταρχάς έχει το λόγο. Γουέντουλιν Ντέλμπος Κόρφιλτ. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ που θα ανεχτείτε ενδεχομένω ε, κάποιες ε, δυσκολίες από πλευρά μου. Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με αυτό το θέμα και θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τους προκατόχους μου που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Είναι ο προπολογισμό λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αφορά το τελευταίο έτος του προηγούμενου πιδελταπή αποτελεί επομένω και τη βάση για το επόμενο πιδελταπή το οποίο θέλουμε να είναι φιλόδοξο ε, και ε, επομένως ε, θα θέλαμε τουλάχιστον μεγαλύτερη φιλοδοξία από ότι η πρόταση της Κομισιόν και κυρίως από τις προβληματικές προτάσεις του Συμβουλίου. να σας πω ποια είναι τα κρίσιμα σημεία. Πρώτον, μείωση του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης Ένταξης. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να ενδυναμωθεί ε, και το θέμα αυτό, καθώς επίσης ε, και το θέμα των, της κατανομής. Θέλουμε αύξηση, βλέπουμε και είναι καλό για τις περιπτώσεις ΔΕΗ. Εδώ έχουμε κάποια αύξηση επίσης 34 4,8% ε, για το 2020 ε, η αύξηση για την ακτοφυλακή και τη συνοριοφυλακή είναι μακράν η μεγαλύτερη αύξηση για τις υπηρεσίες ε, ΔΕΗ. Ελπίζουμε ότι τα χρήματα αυτά, τα αυξημένα, θα χρησιμοποιηθούν για να σωθούν ζωές στην Μεσόγειο και όχι μονάχα για να εμποδίσουμε τους μετανάστες να την περάσουν. Να υπενθυμίσουμε επίσης και τον σημαντικό ρόλο της εισαγγελία για την ε, και επομένως την ανάγκη πόρων πριν από το 2020 έτσι ώστε να είναι λειτουργική ε, η παρουσία. Ε, στο CPD ε, έχουμε μία αύξηση της, ε, ε, της χρηματοδότησης για τον κανονισμό 19 εκατομμύρια για την υλοποίηση του κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ενδεχομένω το ποσό δεν θα είναι αρκετό και θα πρέπει να αυξηθεί. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω τώρα. Εντάχει τα είπαμε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Σκιώδη εισηγητής, σκιώδη εισηγητές μάλλον. Έχουμε πρώτα απ' όλα την κυρία Βόζεμπερκ, η οποία από ό,τι βλέπω θέλει να μιλήσει. Κυρία Βόζεμπερκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι σκιώδη εισηγήτρια. Κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι σκιώδη εισηγήτρια. Ζήτησα το λόγο όταν θα ανοίξετε τον κατάλογο ομιλητών. Μπορώ να μιλήσω τώρα. Δεν είμαι, δεν είμαι shadow. We're replacing the EPP. Δεν αντικαθιστάτε το σκιώδη. Α, Σντεχόφσκι είναι ο σκιώδης του ΕΛΚΑ. Έτσι. Not, not here. Then, if you don't mind, go for the rest of the groups. Τότε ας ακούσουμε τους υπόλοιπους σκιώδης και μετά Εντάξει, συμφωνώ. Ε, σας ευχαριστώ. Ωραία, εντάξει, λέει ο Πρόεδρος. Κρίστιαν Τέρμες, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Thank you. Yes, I'm here. Uh, thank you. Thank you, Chairman. Dear colleagues, as the Σας ευχαριστώ. Εγώ είμαι ο σκιώδης συγκητής για τους σοσιαλιστές, για το όσον αφορά τον προϋπολογισμό, για την ε, χρήση 2020 και ευχαριστούμε τον πράσινο συγκητή για το έργο του. Για τους ε, σοσιαλιστές είμαστε υπέρ των βασικών στοιχείων του σχεδίου του κειμένου, αλλά έχουμε και κάποιες προσθήκες που προτείνουμε, ώστε να αναβαθμίσουμε κάποιες ε, πλευρές του θέματος. Πρώτα-πρώτα, οι πόροι για να έχουμε πιο βιώσιμη πολιτική όσον αφορά διάσωση ε, στην Μεσόγειο. Και όσον αφορά τη θέση των ε, πολιτικών ομάδων για το θέμα της μετάφρασης να μην ξεχνούμε ότι μιλούμε τώρα για ανθρώπους και τα κράτη-μέλη επομένω θα πρέπει να ενθαρρυνθούν για αυτές τις επιχειρήσεις διάσωσης. Επίσης έχουμε εδώ και καιρό στόχο το να βοηθήσουμε την υπηρεσία ασύλου. Ήταν προτεραιότητα το 2016 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να δοθεί κάποια συνέχεια. Επίσης να προσθεθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροφή θα πρέπει να αναβαθμίσει την ε, υποστήριξη προς την ελληνική δημοσιογραφία και τα, την ελευθερία τέλος πάντων των ΜΜΕ. Οπότε να συνεχιστεί η σχετική προσπάθεια, το σχετικό πρόγραμμα, αλλά θα πρέπει οι σχετικές ε, δαπάνες να πάνε προς τα εκεί, προς την ελευθερία του τύπου. Και πάλι να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή και περιμένω την επόμενη συνάντηση, οπότε να δούμε καλύτερα τις λεπτομέρειες με τους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα η κυρία Φαμπιέν Κελέρ για τους φιλελευθέρους έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι μεταφραστές, Ευχαριστώ και την κυρία Γκουίντολίν ε, Κορφίλ Δελμπός για το σημαντικό της έργο και το μεταναστευτικό του 2015 ήταν κάτι σαν ηλεκτροσόκ. Ήταν μια συνειδητοποίηση ότι χρειάζεται περισσότερη συνεργασία, περισσότερη αλληλεγγύη. Και έτσι μπορέσαμε να προχωρήσουμε σε κάποιες σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τις μεταναστευτικές ροές. Και έτσι να προσθέσουμε τα σύνορα και να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη όσον αφορά τους ετούντες άσυλο. Και όπως γνωρίζετε, οι υπηρεσίες της Ένωσης έχουν πολύ σημαντικό ρόλο για αυτή την πολιτική. Βοηθούν τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να υπάρχουν υλικοτεχνικές υποδομές προς τούτο. Πρόκειται για επιχειρησιακές υπηρεσίες. Η γνωμοδότηση νομίζω ότι είναι πολύ καλά ισορροπημένη και καλύπτει την υπηρεσία του ασύλου, την υπηρεσία ε, Frontex, γιατί και οι δύο αυτές οι υπηρεσίες θα έχουν ρόλο κλειδί. Όμως, παρατηρούμε ότι το θέμα της αύξησης πρικοδότησης, της αύξησης του προσωπικού και την ε, Frontex δεν συνάδει με τον ε, στόχο του 10.000 που έχουμε θέσει για το 2027, 2000 ως προσωπικό και επίσης το 2024 που θα προ, κοντά σε αυτό το στόχο. Όπως ελέγχθη επίσης, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το σχετικό ταμείο, το ΑΜΙΦ, όπου έχουμε περικοπή 15%. Αυτά θέλουμε να τονίσουμε για την έκθεση. Επίσης, συμφωνώ με ένα άλλο σημείο. Μας ανησυχεί πολύ. Αφορά τη χρηματοδότηση των δύο αυτών υπηρεσιών. Πρώτα-πρώτα την Ευρωπόλ. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια μικρή αύξηση, αλλά δεν ε, συνάδει αυτό όσον αφορά τα όσα έχουμε πει για την αποστολή της ε, Europol. Είχαμε πει για 35% μέχρι το 2022 όσον αφορά τα νέα μέσα της ε, Europol γιατί γνωρίζετε ότι αυξήθηκαν οι αρμοδιότητες τα τελευταία χρόνια λόγω της Ένωσης για την ασφάλεια, καταπολέμηση της τρομοκρατίας και καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Και πώς θα εξασφαλίσουμε καλύτερη συνεργασία μεταξύ των ε, διοκτικών αγώνων κρατών μελών, εάν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Europol δεν έχει τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους, ώστε να υλοποιήσει αυτή την συνεργασία. Και σας παραπέμπω σε αυτό το 25% του προσωπικού μονίμων υπαλλήλων. Επίσης για μια άλλη υπηρεσία για την οποία είναι ανεπαρκής η Είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι μια καινούργια υπηρεσία που θα πρέπει να αναπτυχθεί για να εκτελέσει την αποστολή της κατά πολέμηση απάτης, όπου και σε αυτό το σημείο θα πρέπει η πρικοδότηση να είναι στο ύψος των φιλοδοξιών. Τέλος. Συμφωνούμε με τις προτεραιότητες για το μεταναστευτικό. Εσείς λέτε βέβαια ότι η αύξηση της ε, προοικοδότησης δεν είναι ε, ανάλογη με το ότι έχουν αυξηθεί μεταστευτικέ ροέ από το 2015 και μετά. Ε, βέβαια όμω είναι απαραίτητο να υπάρχει έλεγχο στα σύνορα και έτσι να μπορέσουμε να προκαταλάβουμε, να προλάβουμε τέλο πάντων την αύξηση των ροών στο μέλλον. Να υπάρχει ασφάλεια στην Ένωση. Είναι προτεραιότητα η πολιτική του ασύλου και ταυτόχρονα θα πρέπει να βελτιώσουμε τη διεκπαιρέωση των αιτήσεων ασύλου, επίσης την υποδοχή των ε, προσφύγων στο μέτωπο της ε, Μεσογείου. Άρα αυτοί οι δύο στόχοι πάνε χέρι-χέρι, μην τους θεωρούμε αντιφατικούς. Πολύ σημαντική και οι δύο αυτοί στόχοι. Τώρα, όσον αφορά τη διεκπαιρέωση των αιτήσεων ασύλου, θα πρέπει το Κοινοβούλιο να ασχοληθεί πολύ με το θέμα να υπάρχει περισσότερη αλληλεγγύη προβασκά των μελών και περισσότερη ασφάλεια για τους πολίτες της ε, Ένωσης αλλά επίση και να προστατευτούν και αυτοί οι οποίοι ζητούν την διεθνή προστασία. Ιωακήμ, από το ECR. Στα πολωνικά. Η κυρία Βυσνιεύσκα. Θα τον αντικαταστήσω εγώ τον Ιωακή. Δεν μπόρεσε να παραστεί Λόγω λοιπόν αυτού του προβλήματο που είχε θα σα ε, πω εγώ την δική του γνώμη. κύριε και κύριοι, ευχαριστούμε τον εισηγητή, την εισηγήτρια τέλο πάντων. Το 2020 ήταν η τελευταία χρήση όσον αφορά το ισχύον ε, πλαίσιο και θα πρέπει επομένως για την αρχή. αυτή να έχουμε πληρωμές στο ίδιο επίπεδο, αλλά να δούμε τι θα γίνει και τα επόμενα χρόνια, να δούμε τι θα γίνει, τόσο ώστε να μην αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των καθυστερήσεων των πληρωμών. Να μην επαναληφθεί το πρόβλημα το οποίο εμφανίστηκε στο παρελθόν. Μιλάμε για 30 δις το 2015. Δεν καταβλήθηκαν αυτά τα χρήματα. Τώρα για το τρίτο κεφάλαιο. Εδώ έχουμε πάνω από 20% των πληρωμών και βέβαια πρέπει κάτι να γίνει για το μεταναστευτικό και για την προστασία των συνόρων μας. Άρα για τον προϋπολογισμό του 20 συμφωνούμε με την αύξηση της πρικοδότησης για τις υπηρεσίες όπως η Frontex. Επίσης, συμφωνούμε με το όργανο ευελιξίας για να καλυφθούν τα υπόλοιπα μέτωπα του τρίτου κεφαλαίου, όπως οι μεταναστευτικές ροές, η ασφάλεια κλπ νέες ανάγκες, νέες προκλήσεις που επιβάλλουν να είναι προτεραιότητα το μεταναστευτικό. Όμως, να είμαστε προσεκτικοί, να μην ξεχνούμε ποια είναι η τάση. Και άρα να προσέξουμε την ευελιξία όσον αφορά τις μεταφορές πόρων πάντα στο, για, για ασφάλεια και μετανάστευση. Θα υποβάλουμε τροπολογίες σχετικά με αυτά. Σα ευχαριστώ. Εκ μέρου τη ΓΚΟΕ. Η Φράου Κορνίλια Έρνστ, λέει ο πρόεδρο. Δεν ξέρω αν είναι εδώ, δεν είναι. Την αντικαθιστά κάποιο. Από την ΚΟΕ υπάρχει κανεί που να είναι πρόθυμο να λάβει το λόγο. Εκπροσωπεί την ΚΟΕ εδώ. Όχι. Άρα πάμε στην ταυτότητα και δημοκρατία ID. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε για τη γνωμοδότηση την εισηγήτρια. Συμφωνώ ε, με την, ε, τον προβληματισμό σχετικά με την μείωση των κονδυλίων για το άσυλο που αντιτίθεται στους ίδιους τους στόχους του ε, Ταμείου. Δεν συμφωνούμε με την ε, κατανομή στους ε, διάφορους, στις διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού, γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βάση σε τις συμφωνίες με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την επανεισδοχή. Προτεραιότητά μας είναι να υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια έτσι ώστε να απαντηθεί ο το πρόβλημα της μετανάστευσης και ε, μέσα από προγράμματα στη στήριξη των χωρών προέλευσης αλλά ε, και ε, με συμφωνίες με χώρες διέλευσης. Όσον αφορά τώρα τις διάφορες υπηρεσίες του χώρου ΔΕΗ, Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε ε, μεγάλη σημασία σε αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες ε, αντιμετωπίζουν και προβλήματα που συνδέονται και με τη μετανάστευση και με την ασφάλεια. Γι' αυτό λοιπόν αντιτιθέμεθα σπόδρα στην μείωση των κονδυλίων της ε, Europol και θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω οι εσωτερικοί μηχανισμοί ασφάλειας όπως η Europol. Επίσης θα πρέπει να ε, υποστηρίξουμε γραμμές ε, οι οποίες ε, θέλουν να αντιμετωπίσουν την ριζοσπαστικοποίηση καθώς επίσης την τρομοκρατία και την, το οργανωμένο έγκλημα. Εμείς θα υποβάλουμε τροπολογίες κατά την έννοια αυτή και ευελπιστώ ότι οι συνάδελφοι θα υποστηρίξουν τις εν λόγω τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Προχωρώ με τους υπόλοιπους ομιτές, τους υπόλοιπους άνθρωπους που έχουν ζητήσει το Βόζεμπεργκ, Τώρα είναι η σειρά σας, κυρία Βόζεμπερκ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να συγχαρούμε την εισηγήτρια και τους συναδέλφους τους σκιώδης εισηγητέ για τις προτάσεις τους. Εγώ θέλω να εστιάσω, για όσους δεν με ξέρουν είμαι Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, από τη Νέα Δημοκρατία, ανήκω στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ε, να πω ότι η χώρα μας, η οποία ανήκει στον Ευρωπαϊκό Νότο, ξέρουμε όλοι ότι έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ από το ζήτημα της μετανάστευσης, η οποία ούτως ή άλλως ε, ως ε, θέμα επιβαρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγιναν πολύ σημαντικά βήματα την πενταετία που πέρασε, παρά τα αυτά το γεγονός ότι οδηγηθήκαμε σε εκλογές. Χωρίς να έχει αναθεωρηθεί το Δουβλίνο, ξέρετε ότι μας το χρέωσαν οι Ευρωπαίοι πολίτες σε όλη την Ευρώπη και είδαμε να αποτυπώνονται αυτές οι χρεώσεις με την αλλαγή της ανθρωπογεωγραφίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρώ ότι το, το ποσό αυτό το μεγάλο που δεν διατέθηκε για την αναθεώρηση του Δοβλίνου, οπωσδήποτε ένα μεγάλο μέρος πρέπει να διατεθεί στο Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, όχι μόνο για τις χώρες που επιβαρύνονται, αλλά για να μπορέσει να βοηθήσει, ούτω ώστε να δούμε περισσότερη αλληλεγγύη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων, σε συνδυασμό με την διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών, αλλά και των προσφύγων μεταναστών είναι κάτι που απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθημερινά δίνουμε εξετάσεις πάνω σε αυτό και σε κάθε περίπτωση οι χώρες που, ε, που επιβαρύνονται περισσότερο ως πρώτες πύλες υποδοχής, όπως είναι η Ελλάδα, είναι εκείνες οι οποίες έχουν περισσότερη ανάγκη. Και τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι αναμφίβολα, πέραν των όποιων ρυθμίσεων κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση του πολύ σοβαρού αυτού θέματος, έχουμε και έναν γείτονα δύσκολο, που από μιλάω για τον Πρόεδρο Ερντογάν, που αντιδρά στις αποφάσεις που εμείς έχουμε πάρει ως Ευρωπαϊκή Ένωση, με απειλή να ανοίξει ανεξέλεγκτα τις πύλες και να γεμίσει την Ευρώπη με απελπισμένους ανθρώπους τη διαχείριση διαχείριση των οποίων δεν θα είναι εύκολο όλες οι χώρες να τη διαχειριστούμε με τρόπο δίκαιο. Έτσι λοιπόν στηρίζω και εγώ ως Ευρωβουλευτής και ως ΕΛΚ τις προτάσεις των εισηγητών οι οποίες είναι κατά το μάλλον ή των συγκλίνουσες στην κατεύθυνση του να ενισχυθεί το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης προς όφελος όχι μόνο των χωρών που πρωτίστως και κυρίως επιβαρύνονται αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εστιάζει στο κράτος δικαίου, στην ελληνική και στις ίσες ευκαιρίε και στι υποχρεώσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Now, Madame Guillaume. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Γκυγιώμα, ευχαριστώ την ε, εισηγήτρια για τη δουλειά της. Ε, πολύ καλά ξεκινάμε. Ε, αν κατάλαβα καλά τα χρήματα που προέρχονταν, μάλλον που θα δίνονταν στη μετεγκατάσταση ε, και δεν χρησιμοποιούν. Μάλλον, να τα ξαναπώ, λέει η ομιλήτρια. Λοιπόν, υπήρχαν κάποια χρήματα τα οποία θα δίνονταν για τη μετάφραση του Δουβλίνου και για το νέο πλαίσιο μετακατάσταση. Και αυτά πήγαν κάπου αλλού. Το καταλαβαίνουμε γιατί αυτή τη στιγμή κάπως έχει τελματώσει κατάσταση με το Δουβλίνο. Και επίσης και το άλλο ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν έχει προχωρήσει ιδιαίτερα pour l'instant de base juridique. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Πώς μπορούμε να έχουμε λοιπόν ε, επαρκείς εγγύησεις για την ε, ε, επαναχρησιμοποίηση αυτών των χρημάτων για τα debarkation mechanism. No. Όταν δηλαδή έχουμε αυτές τις αφήξεις. Προκατσίνη από το ECR. Yes, please. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα μόνο να πω ότι θεωρώ ε, μη ισορροπημένη την προσέγγιση που κάνει η συνάδελφος στη γνωμοδότησή της. Συμμερίζομαι την άποψη βέβαια ότι η μείωση της ε, ε, μάλλον να το πω διαφορετικά λέει ο μιλητής, ε, ότι χρειάζεται οπωσδήποτε ε, κατάλληλη οικονομική κάλυψη της, του επαναπατρισμού, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει το σύστημα των επαναπατρισμών, να γίνει λέω πιο αποτελεσματικό, γιατί αυτή ήταν μια μεγάλη ε, αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το γεγονός επίσης ότι έχουν μειωθεί οι πόροι για την εσωτερική διαχείριση της, ε, του μεταναστευτικού στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να περάσει αλλά παραμένουν θέματα ανοιχτά όσον αφορά την συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και τις χώρες διέλευσης Γι' αυτό, όπως είπε και η Σάνσο Βυσνιέσκα προηγουμένως, εμείς του ECR θα προτείνουμε τροπολογίες έτσι ώστε να ενισχυθεί ε, και ο προϋπολογισμός για την ε, αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και πρόληψη τρομοκρατίας και διαστηνοριακής εγκληματικότητας. Πρόεδρος. Βλέπω ότι όλο και μεγαλώνει ο κατάλογο των ομιλητών και δεν πρέπει να υπερβούμε το χρονοδιαγράμμα μας. Συντέγγι από το ΕΛΚ είναι ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Ήθελα να πω πόσο σημαντικό φυσικά ε, είναι το θέμα του προπολογισμού που έχουμε ενώπιόν μας. Εγώ προσωπικά πιστεύω πως ε, χρειάζονται σαφείς πολιτικές τοποθετήσεις ό,τι αφορά τη μετανάστευση της δυνατότητας της Ευρώπης ε, και επίσης πιο σαφής τρόπος και δυνατότητας προστασίας των Ευρωπαϊκών Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για μεγαλύτερη σταθερότητα και για να δοθεί και ένα τέλος ε, στην κρίση που πολλέ φορέ έχει και ανθρωπιστικό ε, πρόσωπο. Και εξ αυτών ε, συνάγω το συμπέρασμα ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις χρηματοοικονομικέ δυνατότητε, να στηρίξουμε την Ευρωπόλ, τη Eurojust και τη ΕΠΟΛ εν γέννη, να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάτι άλλο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι πω οι μετανάστε που έχουν φτάσει τα τελευταία δύο-τρία χρόνια στην Ένωση αλλά δεν έχουν δικαίωμα παραμονής θα πρέπει να επαναπατριστούν με έφτακτο, ειρηνικό και επαγγελματικό τρόπο. Αυτό πρέπει να γίνει, γιατί αν δεν γίνει, το μόνο που θα πετύχουμε είναι να αυξήσουμε ε, τις ε, παρατυπίες της όλης ε, κατάστασης. Δηλαδή θα ενισχύσουμε το παρά, την παράτυπη μετανάστευση. Έξω και είναι σημαντικό με το σχέδιο περιπολισμού να δώσουμε επαρκή στήριξη στους οργανισμούς και στις πολιτικές που είναι σημαντικές. Μπόλεφα από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και την εισηγήτρια και τους κοιόντες εισηγητές και έχω μια γενική παρατήρηση οποία είναι η εξή. Σε ό,τι αφορά την πολιτική ε, δέσμευση για το gender mainstream, την ισότητα των φύλων, αυτό είναι μια προτεραιότητα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν βλέπω να αντικατοπτρίζεται συνολικά στο σχέδιο προπολογισμού. Το gender budgeting είναι μια μέθοδο που θα έπρεπε να επιτρέπει και σε ό,τι αφορά ειδικέ ανάγκε ανθρώπων και γυναικών να γίνεται η διάκριση και να προβλέπεται χρηματοδότηση. Και το λέω συγκεκριμένα αυτό, διότι σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την κακοποίηση ε, των ε, γυναικών και των κοριτσιών. Και πραγματικά ε, βλέπουμε να υπάρχει μια τάση μείωση των πόρων σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό για το 2020. Το βλέπουμε, αλλά το βλέπουμε και στις συζητήσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και θα πρέπει να το έχουμε όλοι κατά νου το θέμα αυτό, γιατί δεν θέλουμε υποχρηματοδότηση του συγκεκριμένου αυτού τομέα και άλλων ε, σχετικών τομέων. Ο κύριο Παπαδάκη, τώρα, που είναι για έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, το βασικό ζήτημα κατά την εκτίμησή μα δεν είναι μόνο τα ποσά των, τα μεγέθη δηλαδή του προπολογισμού, αλλά το κύριο είναι ο προσανατολισμό αυτού του προπολογισμού και συνολικά της Ευρωπαϊκή Ένωσης που και στο μεταναστευτικό είναι η ενίσχυση της καταστολής, της βάρβαρης καταστολής, των μηχανισμών δίωξης προσφύγων και μεταναστών, μηχανισμών όπως ε, η Europol, ε, η Eurojust, ε, το Ευρωφακέλωμα με όλους τους μηχανισμούς που έχουν διαμορφωθεί, ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή, Ακτοφυλακή και η Ευρωεισαγγελία που αντικαθιστά ακόμα και θεσμούς στα αστικά κράτη. Το κύριο για μας είναι αυτός ο προσανατολισμός, ο αντιδραστικός ε, να ε, ανατραπεί, ακριβώς γιατί αυτό που χρηματοδοτεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο εγκλωβισμός και η συγκέντρωση στα ελληνικά νησιά και σε άλλες πύλες εισόδου ε, προσφύγων και μεταναστών. Αυτό που, αυτό που χρηματοδοτεί είναι να ζουν αυτοί οι άνθρωποι σε άθλιες συνθήκες, σε μόριες, σε απαράδεκτα κολαστήρια των hot spot που τώρα πρέπει να κλείσουν και από αυτή τη σκοπιά αυτός ο προϋπολογισμός ε, συντηρεί, προωθεί και επεκτείνει αυτή την βαρβαρότητα που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια που ανεξάρτητα αν ανεβαίνουν ή μειώνονται οι ε, ροές που σήμερα αυξάνονται ε, το πρόβλημα μένει και συνεχίζεται ακριβώς γιατί η γενεσιουργή αιτία του, η υπεραλιστική πόλεμη είναι παρόντες και έχει ευθύνες και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμμαχή της. Now it's S&D. Κνίτσι. Ευχαριστώ την ε, συνάδελφο, την εισηγήτρια για τη σημαντική έκθεση επαρκής χρηματοδότηση και όλα τα μέτρα τα οποία θα εγκριθούν στα διάφορα μέτωπα σε ευρωπαϊκές πολιτικές είναι πάρα πολύ σημαντικά. Οπότε τονίζω το ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η επαρκής χρηματοδότηση. Κυρίως για την μετανάστευση. Επίσης κάτι άλλο στο οποίο στάθηκαν τόσοι συνάδελφοι που είναι πολύ σημαντικό και χρειάζεται επαρκώς να χρηματοδοτήσουμε τις υπηρεσίες όπως η Eurojust, η Europol και σας τονίζω το ότι οι περικοπές της ε, Europol είναι πάρα πολύ κακό για την υπηρεσία. Έχει υπασχίσει τα τελευταία χρόνια αυτή η υπηρεσία. Τα ξέρουν οι συνάδελφοι της Επιτροπής. Γιατί μιλούμε για καταπολέμηση των πιο σοβαρών εγκλημάτων, για δουλεμπορία, για κακουργήματα οικονομικά. Οπότε θα πρέπει να θεωρηθούν πολύ σημαντικές σχετικές υπηρεσίες και για την ανταλλαγή πληροφοριών, τη διεθνή συνεργασία, που είναι πολύ σημαντικό για την καταπολέμηση τέτοιων εγκλημάτων. Οπότε αυτό σας ξανατονίζω. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε παρκώς αυτές τις υπηρεσίες με ανθρώπινους πόρους και οικονομικούς. Ευχαριστούμε κυρία Κνίτσι. Τώρα, ως συνήθως, αφού ακούσαμε τους συναδέλφους, να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέτε Κιμέντερ, is that the name? Γκμέντερ, Γκμέντερ ονομάζεστε. Γκμέντερ. Yes, hello, good morning and uh, sorry for the complicated name. Καλημέρα. Συμπαθάτε με για το δύσκολο να προφέρετε όνομα. Ετοιμάστηκα για να μιλήσουμε για το 19, αλλά έχουμε και κάτι διαφάνειες για το 20. Καλά. Αν μπορείτε, πηγαίνετε σε αυτές τις διαφάνειες για να συζητήσουμε για το σχέδιο προϋπολογισμού. Εμάς στόχος μας είναι να είναι ισορροπημένοι τα πράγματα, να καλύψουμε όλες τις ανάγκες, αστυνομική συνεργασία, ε, μετανάστευση και προσπαθούμε να προσαρμόσουμε επομένως τα πόσα των κονδυλίων και για το Ταμείο Μετανάστευσης και το διαχείριση των συνόρων προσπαθήσαμε να καλύψουμε τι χρειάζεται και όσον αφορά το ETS. Πολύ σημαντικό στοιχείο θεωρούμε ότι είναι αυτό για τον προπολογισμό. Επίση, ε, ενισχύσαμε το προπολογισμό για τις ε, ευρωπαϊκές υπηρεσίες που έχουν σχέση με την εσωτερική πολιτική και όσον αφορά το προσωπικό και όσον αφορά την ε, εντολή τους που έχει διευρυνθεί επίσης. Προτείναμε και για το 2020 κάποιες αυξήσεις και για το ΣΕΠΟΛ, την Europol, το Ulysses και όλες τις σχετικές υπηρεσίες. Οπότε παρακαλούμε να μας υποστηρίξετε σε αυτή μας την πολιτική ενίσχυση των υπηρεσιών γιατί είδαμε ότι στο Συμβούλιο υπήρξαν προτάσεις περικοπών για το ΆΜΕΦ και εδώ άκουσα τα σχόλιά σας Κοιτάξτε την επόμενη διαφάνεια όπου έχει προταθεί όπως ε, γνωρίζετε ένα ποσό ε, χαμηλότερο κάτω από το ποσό του 2019 αλλά κοντά στα επιθυμητά γιατί το 2019 όμως ξέρετε είχαμε αναβάθμιση το προπολογισμό σχέση με το παρελθόν. Τα 175 είπαμε να καλύψουμε το ΕΚΟ, το μέσω ε, κατεπηγόντων πολιτικών και το εστία. Οπότε είχαμε αύξηση το 19, το 2020 θα συνεχιστεί το πρόγραμμα, αλλά θα γίνει η χρηματοδότησή του με τον τρόπο που θα σας εξηγήσω και θα συνεχιστεί ό,τι προβλέπει ο προϋπολογισμός του 19. Οπότε για το άμεφ Έχουμε τέσσερις στόχους που χρηματοδοτούνται, επιστροφές, αλληλεγγύη, κατάσταση, υποδοχή, άσυλο, κοινωνική ένταξη και μέτρα για την νόμιμη μετανάστευση. Είναι πολύ σημαντικό όλοι αυτοί οι στόχοι του ΆΜΙΦ να καλυφθούν και στην εξωτερική τους διάσταση, γιατί προβλέπεται μια ανάπτυξη δραστηριοτήτων πολύ συγκεκριμένο στοχοθετωμένο στις τρίτες χώρες σε σχέση με τις ε, αναχωρήσεις. Εκεί δηλαδή που επαν... μετεγκαθίστανται τέλο πάντων οι μετανάστες. Όσοι επίσης δεν καλύπτονται από την διεθνή προστασία να μπορούν να επιστρέψουν. Άρα, σκεφτήκαμε πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα στοιχεία και την εξωτερική διάσταση γιατί τα περισσότερα χρήματα για αυτές τις δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν το μέσο εξωτερικής πολιτικής. Επίσης ε, κάποιο άλλο θέμα την άμεση που εκρεμεί. Έχουμε αυτά τα 460 εκατομμύρια βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου. Αυτά είχαν προβλεφθεί και συνεχίζονται το 2020. Και επίσης υπάρχει πρόταση για τον τρέχοντα προϋπολογισμό να υπάρχει ένας μηχανισμός σε σχέση με τα μέτρα αλληλεγγύης και με την κατάσταση. Άρα όλες οι επιλογές είναι εφικτές σύμφωνα με αυτόν τον προϋπολογισμό με την κατάσταση, αλληλεγγύη, με συγκεκριμένες δράσεις. Να βοηθήσουμε τα συνοριακά κράτη-μέλη όπως η Ελλάδα εκεί που είναι οι περισσότερες ε, αφήξεις και οι περισσότεροι μετανάστες παρόντες. Οπότε είπαμε να γίνει αναδιανομή ευθύ αμέσω. Αυτά τα 90 εκατομμύρια τώρα να διανεμηθούν για κάποιες διεθνείς διασυνοριακές διαδικασίες, για κοινωνική ένταξη και για αστυνομική συνεργασία. Οπότε μεταβάλαμε ελαφρώς την πολιτική μας για αυτά τα χρήματα, γιατί φέτος είδαμε ότι αυτά τα χρήματα που πήγανε στο αποθεματικό πήγανε διότι δεν έχει ακόμα εγκριθεί ο σχετικός κανονισμός. Άρα θα πρέπει όπου υπάρχει αυτή η σχετική επιφύλαξη να έρθει από δική σας πλευρά για να διαθέσουμε τους πόρους. Για μπορέσουμε για τις αποβιβάσεις να ολοκληρώσουμε αυτό το οποίο θέλουμε, πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση που σήμερα προβλέπεται γιατί φυσικά αφήξεις υπάρχουν εδώ και καιρό. Γι' αυτό θέλουμε σταθερό επίπεδο πόρων για το 2020 και για τη διοίκηση των και για το ΑΜΙΦ. Αλλά θέλουν να υπάρχουν ε, αυτά τα κονδύλια, όμως λόγω του τι ισχύει για τον κανονισμό του Δουβλίνου ε, διστάζει το Συμβούλιο και θέλει να πάει σε περικοπές. Thank Σας ευχαριστώ κυρία Γκμίντερ. Ολοκληρώθηκε εγκαίρως λοιπόν αυτό το σημείο της μερισιάς διάταξης και απομένει η αναγγελία της προθεσμίας για την κατάσταση τροπολογιών από πλευρά μου και κατάθεση των για το, τροπολογιών για τον ίδιο τον προπολογισμό του 2020. Είναι 27 Αυγούστου, 12 το μεσημέρι. 27 Αυγούστου. Οπότε θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε στις 5 Σεπτεμβρίου της ε, τροπολογής του προπολογισμού σε συνάρτηση με το έργο το οποίο πρέπει να φέρει σε πέραση και Επιτροπή Προπολογισμών. Και για την γνωμοδότηση και για τις τροπολογίες. Λοιπόν, αυτή είναι η πρότασή μας ό,τι αφορά τις προθεσμίες. Κυρία Γκμίντερ. Έχουμε 20 λεπτά στη διάθεσή μας για το επόμενο σημείο της μέσης διάταξης που είναι ακριβώς η παρουσία της μεταφοράς πιστώσεων. 82 εκατομμύρια ευρώ θέλουμε να μεταφερθούν από το αποθεματικό ταμείο του Δουβλίνου στο ΤΑΜΕ ή ΆΜΙΦ στα αγγλικά, που είναι το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης Ένταξης. Θα μας ε, τα πει η κυρία Γκμίντερ, να μας εξηγήσει τους λόγους που ζητείται αυτή η μεταφορά πιστώσεων. Κύριε Γκμίντερ, Διευθύντρια των Ταμείων Μετανάστευσης και Ασφάλειας, θα μας παρουσιάσει για τα επόμενα 10 λεπτά την πρόταση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω το αίτημα αυτό. Θα ήθελα καταρχάς όμως ε, να ε, πω δύο λόγια για τον ε, Γενικό Προϋπολογισμό 2019 που είναι η πρώτη φορά για το νέο κοινοβούλιο που βλέπει αυτό τον προϋπολογισμό. Πολύπλοκος αυτός ο προϋπολογισμός, έξι συνιστώσεις και κατέτος συνολικά στην περίοδο προγραμματισμού έχουμε 2,8 δισεκατομμύρια κατέτος για τα προγράμματα δαπανών. Αναφέραμε το ΤΑΜΕ, υπάρχει και το ΑΕΣΕΦΑ, υπάρχει το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες. Κάποια ζητήματα έρευνα στο μέσα ασφάλεια στο πρόσφατο 2020 και επίσης έχουμε και μέτρα κατά του λαθρεμπορίου ε, ναρκωτικών και την πρόληψη. Έξι αποκεντραμένοι οργανισμοί υπάγονται εδώ. Europol, ε, Frontex ε, και πολλοί άλλοι. Α, δεν μπορούμε να δούμε τις διαφανείς. Εντάξει, αφού υπάρχει τεχνικό πρόβλημα, δεν μπορώ να σας τα διανύμω, θα σας τα στείλω μετά αυτά τα slides. Ε, έρχομαι λοιπόν στον προϋπολογισμό. Για το 2020 σας είπα ότι επιμείναμε και συμφώνησε το Κοινοβούλιο ότι τα 460 εκατομμύρια είχαν μπει στο αποθεματικό. Αυτά τα λεφτά προβλέπονταν για το Δουβλίνο. Είχαμε ζητήσει να έρθει το αποθεματικό αυτό επιβάλαμε για πρώτη φορά, υποβάλαμε αυτό το αίτημα τον Απρίλιο του 19 για Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και κάποια υποστήριξη στο καταπιστευματικό ταμείο. Η πρώτη δόση αποδεσμεύτηκε και ε, ζητούμε τώρα τα 82,8 εκατομμύρια που απομένουν να αποδεσμευθούν ε, για την μετακατάσταση για το 2020 και για άλλα μέτρα υποστήριξης ε, στήριξης της Ελλάδας. Και υπάρχουν και άλλα 7,2 εκατομμύρια για να φτάσουμε στα 90. Αυτά είναι η συμφορά αλληλεγγύης, αν μπορώ να την πω έτσι, ε, για άλλα προγράμματα που είχαμε συμφωνήσει στη συνδιαλλαγή, το Erasmus Plus και τα λοιπά για την Ελλάδα. Τώρα λοιπόν έχουμε 62,8 εκατομμύρια προς την Ελλάδα για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων το 2019 και για τη μεταγκατάσταση έχουμε 20 εκατομμύρια ε, για τη δέσμευση πόρων ε, σε σχέση με το 2020 και τις μελλοντικέ μεταγκαταστάσεις. Τι γίνεται τώρα με το σχέδιο. Καλύπτονται 50.000 άνθρωποι, θα λήξει στις 9 Οκτωβρίου 69% ε, των δεσμεύσεων καλύφθηκαν, οι άνθρωποι αυτοί μετακαταστάθηκαν ε, και τώρα περιμένουμε τα επόμενα βήματα ελπίζοντας ότι θα έχουμε το σχέδιο κανονισμού για τη μεταγκατάσταση και εγώ θα έλεγα να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία ε, δεσμεύσεων από τα κράτη-μέλη, pledging, με στόχο να έχουμε 20.000 επιπλέον. Από αυτούς ε, μπορούμε να καλύψουμε τις 12.000 ε, πρόκειται για επαναχρησιμοποίηση ε, κάποιων πόρων που σχετίζονταν με το ΤΑΜΕ και την ε, μεταγκατάσταση. Άλλαξαν κάποια πράγματα πέρυσι και μπορούν έτσι αυτά τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν για την μεταγκατάσταση και ήδη έχουν προταθεί 12.000 τέτοιου είδους μεταγκαταστάσεις και Άλλες 2.000 για να έχουμε 14.000 συνολικά θα θέλαμε να τις καλύψουμε από το αποθεματικό αυτό. Ελπίζω λοιπόν να συμφωνήσετε να έρθει το αποθεματικό για αυτή τη δραστηριότητα και οποιαδήποτε άλλη πρόταση θα έχουμε θα προσπαθήσουμε να τη χρηματοδοτήσουμε από τις ε, πιστώσεις ε, του 2020. Αν πάμε τώρα στις δραστηριότητες στην Ελλάδα, 62,5 68,2 εκατομμύρια. σα δώσω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα του τι χρηματοδοτούμε στην Ελλάδα. Χρηματοδοτούμε, όπως είπα, το πρόγραμμα ε, Εστία για την ε, παροχή καταλήμματος ε, στους πρόσφυγες και κάποια μετρητά 120 ευρώ το μήνα παίρνουν οι μετανάστες. Τα διαχειρίζεται η πατερμοστία τους πρόσφυγες αυτή τη στιγμή έχει χρήματα για 70.000 άτομα και θα θέλαμε να μπορέσουμε να αυξήσουμε αυτό το ποσό διότι αφήξει, όπως υπόθηκε από τους βουλευτές αυξάνουν ε, και θα έπρεπε τώρα να είμαστε σε θέση να καλύψουμε 87.000 ε, σε αυτό το πρόγραμμα εστία και ακριβώς λόγω των πολλών αφήξεων πρέπει να φιλοξενηθούν κάποιοι σε ξενοδοχεία. Δεν είναι βέβαια η καλύτερη δυνατή λύση, είναι πολύ δαπανηρή και η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται σκληρά ώστε να υπάρχουν και άλλε δυνατότητε, να υπάρχουν κάποιοι άλλοι ε, χώροι υποδοχή, ε, κάποιοι είδου καταβλισμοί που είναι μια πιο αποτελεσματική λύση, αλλά δεν υπάρχουν επαρκεί ε, εγκαταστάσει τέτοιε προ το παρόν. Άρα προ το παρόν θα χρειαστεί να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε αυτό το έκτακτο σχέδιο μέχρι τον Νοέμβριο. Θέλουμε λοιπόν αυτά τα επιπλέον χρήματα, το οποίο είπα, ε, που είναι 28,3 εκατομμύρια και σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Μετανάστευση. Έχουμε κάποια ως καταβλισμού στην ενδοχώρα. Εκεί χρειάζονται μεταφραστικές υπηρεσίες, διερμηνία, στα σχολεία χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη για τους μετανάστες ε, και τους πρόσφυγες. Χρειάζεται επίσης ε, ε, μεταφορά του προσωπικού και των μεταναστών, εφόσον πολλές φορές αυτοί οι καταβλισμοί βρίσκονται σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές και τα συνόδευτα παιδιά. θέλουμε ασφαλής τοποθεσίες για αυτούς και επίσης επιπλέον ειδικευμένες υπηρεσίες για αυτούς τους ανηλίκους. Ελπίζω να μπορέσετε να αποδεσμεύσετε αυτά τα ποσά, να εγκρίνετε δηλαδή αυτή η μεταφορά, γιατί είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να αποδεσμεύσουμε τα χρήματα αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Γενική Διεύθυνση ε, για τα όσα μας είπε. Ε, Βλέπω ότι κάποια μέλη ζητούν ε, το λόγο. Δεν βλέπω καλά τα ονόματα, λέει ο πρόεδρος. Βλέπω και αναπληρωτές που ζητούν το λόγο. The floor to you, and then it'll be you. Please. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και για την πρωτοβουλία. Έχω περάσει αρκετό χρόνο στα ελληνικά νησιά και η κατάσταση αυτή ε, πραγματικά δεν είναι βιώσιμη και καλό θα ήταν να ε, επενδυθούν ε, περισσότερα χρήματα. Η λογική κυβέρνηση θέλει όχι μόνο να βελτιώσει την κατάσταση του καταβλισμού και να έχουμε περισσότερα θέσει εκεί, αλλά πρέπει να δούμε ότι η χωρητικότητα στα νησιά ε, έχει διευρυνθεί, έχει μεγαλώσει, αλλά και πρέπει ακόμη να διευρυνθεί. Και επίσης, αν μπορούμε να αποκλείσουμε τότε αυτά τα χρήματα, αυτά τα 82 και κάτι εκατομμύρια, ε, να μην επενδυθούν, επαναλαμβάνω να φροντίσουμε να μην επενδυθούν για τη δημιουργία κλειστών κέντρων κράτησης στα ελληνικά νησιά, διότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα κυκλοφορίας ε, και διακίνηση είναι πολλοί αυτοί που δεν μπορούν να, να ε, τους, ε, δεν μπορούν να βγουν καν από αυτά τα κέντρα και πραγματικά θέλω να μας εγγυηθείτε ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν, τέλος πάντων να φροντίσουμε ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν ώστε να δημιουργηθούν κλειστά τέτοια κέντρα. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω ποιο είναι το όνομά σας, αλλά έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Λέγομαι Κώστα Αρβανίτης, είμαι από την Ελλάδα, είμαι από το ΣΥΡΙΖΑ και εκπροσωπώ την ΚΟΕ. Έχουμε τρεις παρατηρήσεις, έχω τρεις παρατηρήσεις να κάνω και θα ήθελα να τονίσω στο σώμα ότι στην Ελλάδα έχουμε αλλαγή κυβέρνησης και έχουμε και αλλαγή δόγματος. Έχουν περάσει τρία χρόνια καταρχήν και τρει μήνε από την έναρξη των συζητήσεων για την αναθεώρηση του κανονισμού του Δοβλίνου για ένα πιο δίκαιο, πιο βιώσιμο σύστημα κατανομή των ετούντων άσυλο. Α, θέλω να συμπληρώσω εδώ ότι το επάγγελμά μου είναι δημοσιογράφο. Έχω περάσει, έχω κάνει χιλιάδε χιλιόμετρα, έχω κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ στι δομέ και στην κατάσταση το πώ, το τι επικρατεί χρόνια τώρα στην περιοχή. Οπότε έχω μια γνώση βιωματική. Ήθελα λοιπόν να σημειώσω ότι δίκαιο για αυτού του ανθρώπου, δίκαιο για τα κράτη-μέλη που του υποδέχονται, δίκαιο για του ετούντε άσυλο, δεν είναι οι αριθμοί. Είναι οι άνθρωποι που χρήζουν διεθνού προστασία, είναι οι αριθμοί, αριθμοί είναι μάλλον είναι τα στοιχεία του μεγέθου του Πλούτου και τη δυνατότητα απορρόφησης του κάθε κράτου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτού του αριθμού σχετίζονται μόνο η έννοια του βιώσιμου. Μα βρίσκει αντίθετου να βλέπουμε με αυτή την οπτική το θέμα. Και φυσικά σημειώνω και σε αυτό που λέει ο κ. Παπαδάκη θα συμφωνήσω ότι βασικό ζήτημα είναι και η αιτία που δημιουργεί προσφυγική κρίση. Ο πόλεμο δηλαδή. Ρωτώ λοιπόν γιατί δεν έχει προχωρήσει αυτή η ζήτηση και για να μπω ακριβώ στο θέμα. Σε ό,τι αφορά στα κονδύλια που συζητάμε. Προφανώ υπάρχει ανάγκη χρημάτων. Προφανώ. Όμω το ζήτημα είναι του πόθεν προέρχονται αυτά τα χρήματα είναι μικρότερη σημασία συγκριτικά με το πού καταλήγουν αυτά τα χρήματα είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε το μηχανισμό που θα αξιοποιήσει η Επιτροπή ώστε να παρακολουθήσει την πορεία αυτών των κονδυλίων. Πώ λοιπόν θα διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα αυτά θα δαπανηθούν για να καλυφθούν οι ανάγκε των ανθρώπων που αιτούνται άσυλο, ότι θα δαπανηθούν στι δομέ που προσφέρουν πραγματικά χρήσιμε υπηρεσίε, ότι θα κατευθυνθούν στην ένταξη και όχι στην απομόνωση, στην επανένωση δηλαδή των οικογενειών και όχι σε fast track επαναπατρίσει, στην περίθαλψη και όχι στη δημιουργία κέντρων κράτηση. Να σημειώσω κάτι, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Όταν είπα στην αρχή άλλαξαμε κυβέρνηση, αλλάξαμε δόγμα, στην Ελλάδα το Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτική καταργήθηκε. Έγινε υπηρεσία στο Υπουργείο Δημόσια Τάξη. Το θέμα για την κυβέρνηση δεξιά είναι αστυνομικό. Δεν είναι όπω το βλέπουν οι περισσότεροι από εμά. Γι' αυτό επιμένω στο κομμάτι αυτό. Πάρα πολύ σημαντικά να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κλείνοντας, στην πραγματικότητα το Υπουργείο του Πολίτη, Προστασία του Πολίτη, επιφορτισμένο με τον έλεγχο και την καταστολή ω κύρια αρμοδιότητα, κατάπιε, όπω σα είπα, ένα ολόκληρο Υπουργείο Μετανάστευση εξαιτία των πολεμικών αιστειών και τη φτώχεια ω ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμεί δεν το βλέπουμε έτσι το θέμα. Με άλλα λόγια, και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, να, προγραμμα... να προπαγανδίσει καταρχά και να διαχειριστεί κατόπιν την αντίληψη ότι οι μετανάστε δεν είναι άνθρωποι ξεριζωμένοι, από τι πατρίδε, κατατρεγμένοι, υποταγμένοι δικαιωματικά στην ομπρέλα προστασία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΙΕ και του Διεθνού Οργανισμού Μετανάστευση. Οι άνθρωποι αυτοί, τέλο, για τη Νέα Δημοκρατία, για τη δεξιά, για το Λαϊκό Κόμμα, είναι ανεπιθύμητοι, όπω το καταλαβαίνω, επικίνδυνοι, μιαρή εισβολή. Ειλικρινά δεν θα μπορούσα να σκεφτώ άλλον τρόπο ώστε αυτή η πρόθεση τη ελληνική κυβέρνηση να γίνει περισσότερο σαφή. Το βασικό ερώτημα είναι, μπορεί η μπορεί τα όργανά μας και με ποιον τρόπο να διασφαλίζει ότι τα χρήματα αυτά να πάνε, αλλά θα πάνε σε υπηρεσίε και όχι σε εγκλισμό και τέτοιες λογική που σας ανέφερα πριν. Σας ευχαριστώ. Thank you, Mr. Avernidis. I saw... De vous, uh, dire... Keller, de Aldi. Vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier... Κυρία Κέλλερ, από τους φιλελευθέρους ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, αλλά και την Επιτροπή που μα έστειλε την εκπροσωπό για την σχετική παρουσίαση και εμείς θέλουμε ε, να συμφωνήσουμε ότι θα πρέπει να δοθούν περισσότερα μέσα επιχειρησιακά για να πλαισιωθεί η προσπάθεια για τους μετανάστες στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς, όπως και άλλοι συνάδελφοι, ε, δεν θέλουμε αυτό να γίνεται μια μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό του Δουβλίνου. Είναι το πιο ρεαλιστικό βέβαια το να χρησιμοποιηθούν κάπου αυτοί οι πόροι. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τι δημοσιονομικέ πολιτικέ του 2020 και έτσι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για μια ευρωπαϊκή στρατηγική. Επίση, ε, κυρία Γκμίντερ, θέλω να σα ρωτήσω για κάτι άλλο. Τι γίνεται με ένα άλλο σημείο αφήξεων, το Γιβραλτάρ, από τη Βόρεια Αφρική προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν προτείνεται μεταφορά πιστώσεων σε σχέση με αυτό. Μπορείτε να μας πείτε τι ισχύει και για το 19 και αλλά και για το 20 και Σαφαλέχο. Αλλά representante de la Comisión. Ευχαριστούμε την Γοσβολή κύριος Θαρθαλέχος. Το πρόγραμμα αυτό οξύνεται συνέχεια. Ε, γίνεται το πρόβλημα των ασυνοδεύτων ανηλίκων. Και αυτό γίνεται παντού στην Ευρώπη και στην ε, Ισπανία, ε, στις ε, πόλεις που συνορεύουν με το Μαρόκο, τις αυτόνομες σχετικές περιοχές, αλλά και σε, σε μεγάλες πόλεις. Θα πρέπει επομένω κάτι να γίνει για βοήθεια, κάπως να διεκπεριώνεται, να διαχειρίζεται η κατάσταση, γιατί πρόκειται για μια κοινωνική ομάδα που είναι πάρα πολύ ευάλωτη όσον αφορά την εκμετάλλευση. Εργασιακή, σεξουαλική. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά και συμβαίνει πολύ συχνά να καταλήξουν σε κάποιες οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες των πόλεων. Και επίσης θέλω να σας πω ότι το πρόβλημα συνεχώς παροξύνεται. Άρα χρειάζεται στοχευμένη δράση, οικονομική πλαισίωση στις σχετικές πολιτικές για βοήθεια στις χώρες που αυτές είναι οι χώρες που καταλήγουν αυτοί οι μετανάστες. Ευχαριστώ για το ΕΛΚΟ κύριο Σόιντο. Ευχαριστώ και εγώ τα όσα μας είπε η εκπρόσωπο της Επιτροπής. Να σας πω δύο σκέψεις μου. Πρώτα-πρώτα να σας πω ότι συμφορώ με αυτή τη ε, μεταφορά των 82 εκατομμύριων ευρώ από το αποθεματικό στο ΤΑΜΕ, στο ΑΜΗΝ, ούτως ώστε να βοηθήσουμε τις ελληνικές προσπάθειες για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα υπάρχουν οι εγγυήσεις σωστής και στα επίπεδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση διεκπαιρέωση των αιτήσεων ασύλου για να δούμε τι θα γίνει σε περιφερειακό τοπικό επίπεδο με του μετανάστε και έτσι να είναι αποτελεσματικά τα προγράμματα για την, για την επιστροφή των επαναπατρισμών. Επίση, να καλύψουν και κάποια πιο συγκεκριμένα ζητήματα, αυτά που τα έθιξε ο συνάδελφο πριν από λίγο. Να λάβουμε υπόψη επίση τι ειδικέ συνθήκε που περιβάλλουν ε, την ε, Μεσόγειο ε, ενώ το Γιβραλτάρ και γενικότερα τις ισπανικές ακτές ε, εν κατακλείδη, μια που έχω τον λόγο, να σας πω και το εξής. Το Συμβούλιο να συμφωνήσει όσον αφορά το τι θα γίνει με τον κανονισμό του Δουβλίνου. Να βρεθεί μια βιώσιμη λύση όσον αφορά την κατανομή των ετούντων άσυλο. Πιο δίκαιη η κατανομή ευθυνών ε, μεταξύ των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σόιδο. Θα δώσω ξανά το λόγο στην κυρία Κμίντερ από την Κομισιόν. Μπορείτε να κάνετε κάποιες τελικές ε, παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και όλους για τα σχόλια. Όντως, ε, όπως ορθώς ε, είπατε, η μη έγκριση ακριβώς ε, και μη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου ε, έχει από την άλλη πλευρά ε, την το αποτέλεσμα, ας πούμε, κάποιες χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να πρέπει να υποδεχθούν μεγάλο αριθμό μεταναστών και επομένως να χρήζουν της βοήθειάς μας. Πρέπει να πω βέβαια ότι εάν συμφωνηθεί το Δουβλίνο, ε, τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν απευθείας για το σκοπό αυτό. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Όσον αφορά τις ερωτήσεις στον κύριο Μάρκο μπορώ να πω ότι οτιδήποτε χρηματοδοτείτε θα πρέπει να σέβεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Επομένως, νομοθεσίες ε, ε, και ε, αρχές τις οποίες έχετε ήδη εγκρίνει θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται σεβαστές. Αυτό είναι εκ των ουκάνευ και οπωσδήποτε δεν μπορεί να υπάρξει καμία χρηματοδότηση με τρόπο διαφορετικό ή με συνθήκες διαφορετικές. Είναι γεγονός ε, ότι και στην Ελλάδα έχουμε δει μεγάλη αύξηση ε, των ε, αφήξεων και ναι, αυτή οδήγησε και σε αύξηση των hot spots και εμείς ε, υποστηρίζουμε ε, την δραστηριότητα αυτή, υποστηρίζουμε να φεύγουν οι άνθρωποι από τα hot spot. Είναι γεγονός ότι τώρα πηγαίνουν σε άλλες ε, δομές και εμείς υποστηρίζουμε την κίνηση αυτή. από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιες ε, δραστηριότητες τις οποίες ε, υποστηρίζουμε ε, εμείς άμεσα τις ελληνικές αρχές όπως ας πούμε όλες οι διαδικασίες για την έφεση. Τα υπόλοιπα χρήματα κανονικά πηγαίνουν σε οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς. Εμείς έχουμε επίσης υπογραμμίσει ότι ε, θέλουμε οπωσδήποτε ιδιαίτερη ε, προσοχή να δίνεται στους ε, ασυνόδευτους ανηλίκους και γι' αυτό υπάρχει και ειδική χρηματοδότηση και έχει δοθεί και ειδική χρηματοδότηση και για την ταυτοποίηση ε, στα κέντρα των, στην Ελλάδα των ε, ανηλίκων που είναι ασυνόδευτοι. Όσον αφορά την Ισπανία τώρα, βρισκόμαστε σε διαδικασία να δώσουμε περισσότερα ε, επιπλέον χρήματα σε projects τα οποία αφορούν την ίδρυση πρόσκαιρων δομών για τους λόγους της ταυτοποίησης των αφικνιωμένων καθώς επίσης ε, και για την δημιουργία κέντρων επίγουσας ε, υποδοχής, ε, βεβαίως και για την χρηματοδότηση της χρήσης επιπλέον δυνάμεων της Guardia Civil που εμπλέκονται στις διαδικασίες αυτές. Αυτό προβλέπεται για αργότερα, δεν το έχουμε, γι' αυτό δεν το ανέφερα σήμερα. Επίσης, όσον αφορά αυτήν, αυτόν τον προϋπολογισμό για frontline support. Ε, έχουμε δώσει χρήματα τα προηγούμενα χρόνια και στην Ιταλία ε, και επίσης ε, συζητούμε και με την Ιταλική κυβέρνηση για προγράμματα τα οποία κυρίως θα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της εργασιακής εκμετάλλευσης κυρίως σε γενικές ε, γραμμές πρέπει να πω ότι τα χρήματα αυτά ε, δίνονται για έναν καλό σκοπό ε, και βεβαίως ότι δίνονται στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, ε, δίνονται σε διεθνείς ε, οργανώσεις ε, και στις εμπλεκόμενες χώρες. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε και μια γενική συζήτηση για τον προσανατολισμό του προϋπολογισμού, για το τι κάνει ο προϋπολογισμός κλπ. Αλλά πρέπει να σας πω ότι μονάχα ε, ένα 30% ε, που αφορά την μετανάστευση ε, το διαχειρίζεται άμεσα η Κομισιόν, η υπόλοιπη διαχείριση γίνεται από τα κράτη-μέλη. Αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μίντερ. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εμπεριστατωμένη εντελεχή αυτή παρουσίαση. σε ό,τι αφορά τη μεταφορά πίστοση ύψους 82 εκατομμυρίων ευρώ. Άκουσα τις παρεμβάσεις των συναδέλφων και ορισμένοι μίλησαν για την ανάγκη απεμπλοκής της κατάστασης με τον κανονισμό του Δουβλίνου. Και θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο από αυτού για να προσπαθώ να εξηγήσω κάπως τα πράγματα. Είχα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων την Πέμπτη και Παρασκευή που μας πέρασε, ε, επί Φινλανδικής Προεδρίας, στο Ελσίνκι λοιπόν. και εκπροσώπησα την υποτροπή μας, ε, από την ιδιότητά μου Προέδρου της, ως ήθιστε, και φυσικά πήρα και το λόγο στη συγκεκριμένη αυτή συζήτηση για το μέλλον της μεταναστευτικής πολιτικής. Αυτό ήταν το θέμα. Σε αυτό το Συμβουλίο Δικαιοσύνη Εσωτερικών, το ΔΕΗ, έκανε κάποια σχόλια η Φιλανδική Προεδρία στο Ελσίνη και μίλησε για την εσωτερική ασφάλεια, την τεχνητή νοημοσύνη, τι υβριδικέ απειλέ, την ενίσχυση του κράτου δικαίου και τη δικαστική συνεργασία σε ποινικά θέματα. που είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα όπως καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε. Και υπόθηκε ξεκάθαρα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ζητά και θέλει το στόματρο δυνατό να δοθεί εντολή στη Φλαδική Προεδρία για να ξεκινήσει ε, διαπραγματεύσει που θα οδηγήσουν σε άρση του αδιεξόδου για το Δουβλίνο, ώστε να μπορέσει να ξεπλοκαριστεί όλο το πακέτο για το άσυλο, διότι υπάρχουν ε, κρεμή ζητήματα που είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ του. Ο κανονισμό Eurodac, για παράδειγμα. Όλα αυτά έχουν μπλοκαριστεί. Το είπα και ξεκάθαρα επομένω το δήλωσα. Όλα αυτά έπρεπε να είχαν εγκριθεί όχι σήμερα, πριν από χρόνια. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Έχουν μπλοκαριστεί όλοι αυτοί οι κανονισμοί λόγω το ότι δεν υπάρχει κοινή θέση και συμφωνία σε επίπεδο συμβουλίου σε ό,τι αφορά το Δουβλίνο. Και σε αυτό το Συμβούλιο ΔΕΗ στη Φιλανδία, δικαιοσύνη εσωτερικών υποθέσεων, έγινε μια θερμό συζήτηση, παρουσία του Επιτρόπου Αβραμόπουλου που έθεσε και το θέμα των αποβιβάσεων και τις ε, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. Σε ό,τι αφορά ε, την έλλειψη συμφωνίας ε, επανεισδοχής, δεν ξέρω μήπως θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί το θέμα των θεωρήσεων διαβατηρίου απελευθέρωση το καθεστώτος αυτού. Εγκρίθηκε ο κώδικας θεωρήσεων ε, στο τέλος ε, της προηγούμενης θητείας. Και ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκε είναι η εμπορική πολιτική. Υποχρεωτικές ε, διαδικασίες στα σύνορα και πολύ καλή ανάλυση και εξέταση για να μπορούμε να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης αφενός και διακίνηση αφετέρου, εμπορίας ανθρώπων δηλαδή. και σχετική ε, οδηγία έχουμε στις πολλές φορές να τροποποιηθεί. Συζητήθηκε επίσης ο κατάλογος των ασφαλών τρίτων χωρών. Ειδήσει για τις βόρειες ακτές Αφρικής και Λιβύη ήταν το συγκεκριμένο, το πιο συγκεκριμένο θέμα που ετέθη οι υπουργοί και συγκεκριμένα ο αρμόδιος φυλαδός θα έρθει εδώ αρχές Σεπτεμβρίου, 4 Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά τις θερινές διακοπές θα έχουμε την ακρόαση με τον αρμόδιο φυλαδό υπουργό για αυτά τα θέματα. Για να σας πω ότι αυτά τα συζητήσαμε και μάλιστα ενδελεχώς ε, ευκαιρία του Συμβουλίου Δικαιοσύνης Εσωτερικών Υποθέσεων που έγινε στην αρχή της ανάληψη της Φιλανδική Προεδρίας. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι το σημείο 5 ή 6 στη Μέση Διάταξη. Θα κάνουμε ένα fitness check, έναν έλεγχο καταλληλότητας, έτσι το λέμε. Έχουμε μια ώρα γι' αυτό. Και εδώ συζητούμε την νόμιμη μετανάστευση. Το Μάιο 2015 είχε δημοσιευτεί το θεματολόγιο της Κομισιόν και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχει λήξει και να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2018. Όμως, τι έγινε στην προηγούμενη θητεία. Δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας και δεν κλείσαμε το φάκελο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, έχουμε αυτό το θέμα σήμερα στη μέση διάταξη για να συζητήσουμε τρεις συγκεκριμένα οδηγίες ε, την υλοποίηση τριών οδηγιών. Την οδηγία του 2003 σε ό,τι αφορά την νόμη μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, την οδηγία του 2003 σε σχέση με το καθεστώς υπηκών τρίτων κρατών που είναι επιμακρών διαμένοντες. Επίσης, δεύτερο, οδηγία του 2003 για το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση και τρίτον, την οδηγία του 2011 για την ενιαία άδεια σε επικοστρίτων των κρατών. Εκεί θεσπίζονται δικαιώματα, μια κοινή δέσμη δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος. Πριν από 20 χρόνια στο Τάμπερε είχε παρουσιαστεί από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εξωτερικών ένα εγγράφω κάποια απορίσματα, 20 χρόνια πριν επαναλαμβάνω, ε, σε σχέση με τους αλλοδαπούς εργαζομένους. Τα τελευταία χρόνια, όπως όλοι γνωρίζουμε, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν εντοπίζεται πλέον ε, συγκεκριμένα σε όλους τους εργότες, αλλά κοιτά κυρίως το, σε εποχιακούς εργαζόμενους, ενδομιλικές αποσπάσεις, ε, φοιτητές, ε, ερευνητές. Νομίζω ότι είναι καιρός πλέον να δούμε πιο οριζόντια τα πράγματα μέσω των τριών αυτών οδηγιών τις οποίες προανέφερα. So far, in which... Χρειάζονται βελτιώσεις, αυτό είναι σαφές. Έχοντας όλα αυτά υπόψη για την νόμιμη μετανάστευση, θα δώσω το λόγο στον κύριο Ματίας Ελ, που είναι Διευθυντής Μετανάστευσης ε, Κινητικότητας και Ενοτομίας. Θα έχετε εσείς κύριε Έλ το λόγο και στη συνεχεία θα ακολουθήσετε τα λίγα Παρακαλώ. Thank you very much, Mr. Mr. Chairman, and uh, this is my. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι η πρώτη μου φορά ε, στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή σας και γι' αυτό θα ήθελα να σας πω και επισήμως ότι πραγματικά προσδοκώ ε, καλή συνεργασία με το νεοεκλεγέν ε, σώμα την 1η Απριλίου, κυρία Πρόεδρε, μετά από την δημοσιοποίηση του ε, γράφου εργασίας της Κομισιόν για τον ε, έλεγχο καταλληλότητας. Ε, είχαμε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ξεκίνησε η συζήτηση και τώρα θα παρουσιάσουμε τα κύρια συμπεράσματα των κύριων ε, οδηγιών για τη μετανάστευση που αναφέρατε είναι μερικοί νέοι εδώ στο Κοινοβούλιο και δεν γνωρίζουν καλά τα, την αλληλουχία. Γι' αυτό θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις όσον αφορά τον έλεγχο καταλληλότητας και τα όσα έχουν συμβεί από τον Απρίλιο. Ε, πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσω ότι τα αποτελέσματα του fitness check απέδειξαν ότι είναι σημαντικό να έχουμε πολιτική νόμιμης μετανάστευσης που θα πρέπει να αποτελέσει κεντρικό στοιχείο της ε, ε, ε, αντιμετώπισης που θα έχουν τα μεταναστευτικά ρεύματα από την Ευρώπη. Δηλαδή η νόμιμη μετανάστευση είναι αποτελεσματικός ακρογωνιαίος λήθος για την γενικότερη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το fitness check ε, κατέδειξε ότι υπάρχουν ήδη θετικά στοιχεία όσον αφορά τη διαχείριση νόμος μετανάστευσης. Ας πούμε, ε, έχουν αυξηθεί τα δικαιώματα των νομίμως διαμενών των ε, πολιτών τρίτων ε, χωρών ε, και έχει βελτιωθεί και η διαδικασία οικογενειακής ε, επανένωσης ενώ υπάρχουν άλλα στοιχεία τα οποία δεν έχουν στεφθεί από μεγάλη επιτυχία. Ε, ας πούμε δεν υπάρχει αρκετή θελκτικότητα, ελκυστικότητα όσον αφορά ε, δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες ε, και επομένως και όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε έχουμε και κάποια προβλήματα υλοποίησης το σημαντικό είναι να προετοιμάσουμε καλά το έδαφος για την επόμενη ε, Επιτροπή. Γι' αυτό και την 1η Απριλίου ε, ε, και ένθεν έγιναν πολλές στοχευμένες συζητήσεις και επαφές με εθνικούς εκπροσώπους που πρέπει να σας πω ότι επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει ανάγκη ενωσιακής νομοθεσίας που θα εστιάζει στις κατηγορίες ε, των εργαζομένων και των προσώπων που ε, χρειάζονται κατηγοριών εργαζομένων που χρειάζονται περισσότερο. Μη κυβερνητικέ οργανώσεις και συνδικάτα ζητούν καλύτερους ε, κανόνες για την οικογενειακή επανένωση, καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των μεταναστών. Ε, ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες επίσης ε, υπογραμμίζουν ότι θα πρέπει ναι να υποστηρίξουμε ε, την έλευση λιγότερο εργαζομένων με λιγότερα προσόντα, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να προσεγγίσουμε και ανθρώπους με συγκεκριμένο προφίλ όπως κάνει η Αυστραλία. Ε, Γενικώ ε, υπάρχει ανάγκη στοχευμένης καλύτερης βελτίωσης ε, του υπάρχοντος πλαισίου παρά η δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου και έχει υπάρξει συμφωνία ότι ναι, έχουμε δει προόδους και θα πρέπει να επικεντρώσουμε στην περαιτέρω βελτίωση. πρέπει να προταθούν συγκεκριμένα στοχευμένα νομοθετικά ε, μέτρα. Επί τη βάση όλων αυτών, κύριε Πρόεδρε, εμείς ε, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη, προτιθέμεθα δηλαδή να λάβουμε σοβαρά υπόψη τα αποτελέσματα αυτής της ε, διαβούλευσης και πολιτικά θα πρέπει να συζητήσει η επόμενη Επιτροπή για το πώς θα κινηθεί στο θέμα της μετανάστευσης. Όσον αφορά τώρα τα συμπεράσματα του Implementation Report ε, για την ε, ε, ενιαία άδεια παραμονής και την οικογενειακή επανένωση. Σε αυτά να πω κάποια γενικά πρώτα είναι υποχρέωση η έγκριση μιας τέτοιας έκθεσης. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Είναι ε, υποχρέωση να υπάρχουν τέτοιες εκθέσεις. Δεύτερον, η ανάθεση της, ε, η υποχρέωση μάλλον ε, της ε, παρακολούθησης της υφιστάμενης νομοθεσίας καθώς επίσης και η πρόταση για νέα νομοθεσία αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, κατά την έννοια αυτή λαμβάνονται υπόψη είναι και οι εθνικές προσεγγίσεις όσον αφορά την οδηγία για την οικογενειακή επανένωση ε, επιβεβαιώνεται στην έκθεση ότι η υλοποίηση έχει βελτιωθεί ε, έχουν ξεκινήσει και διαδικασίες επί παραβάση από την Κομισιόν, αλλά έχει συμβάλει σε αυτό ε, και ε, η διδράση της Κομισιόν που ξεκίνησε το 2004, καθώς επίσης και κάποιες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υπάρχουν παρόλα αυτά και ταυτοποιούνται ε, και αναφέρονται στην έκθεση πολλές προκλήσεις όσον αφορά ας πούμε την επιβεβαίωση των ταυτοτήτων των ε, μελών της οικογένειας που αποτελεί διαδικασία ε, μακρόχρονη ε, και απαιτεί πολύ μεγάλους χρόνους. Όσον αφορά τώρα την οδηγία για την μακρά παραμονή, ε, στη βελτίωση της κατάστασης έχουν συμβάλει και κινήσεις της Κομισιόν και αποφάσεις του δικαστηρίου. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία ε, δυναμητίζουν την υλοποίηση των κύριων στόχων της ε, οδηγίας υπάρχουν χώρες ας πούμε οι οποίες δεν έχουν ακολουθήσει το σύστημα ε, των αδειών μακράς ε, παραμονής και επιμένουν στα εθνικά, στις εθνικές άδειες ε, παραμονής. Υπολείπονται λοιπόν τα ευρωπαϊκά σχήματα. μονάχα 3,1 εκατομμύρια ε, υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν αυτή την ευρωπαϊκή άδεια ε, σε αντιπαράθεση με 7 και πλέον εκατομμύρια που έχουν εθνικές άδειες παραμονής. Ε, όσον αφορά τώρα το κεκτημένο και τα ειδικά, τις ειδικές διατάξεις, να πούμε ότι η πρώτη έκθεση υλοποίησης ε, αναφέρεται ε, σε κάποια προβλήματα, κυρίως σε σχέση με τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Ε, τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, εάν πρέπει να αναπτυχθεί η, και προς τα πού πρέπει να αναπτυχθεί η ε, μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα αποφασιστεί από την Κομισιόν και τους ε, νομοθέτες. Ε, η νομική βάση που υπάρχει αποτελεί ήδη μια ικανή νομική βάση. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνουν πολιτικές συζητήσεις και θα πρέπει ε, οι ε, οδηγίες να εφαρμοστούν σωστά σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει δε και η ανάγκη βελτίωσης των πληροφοριών που διατίθενται στους, στις τρίτες χώρες και στους υπηκόους τρίτων χωρών που προτίθενται να μετακινηθούν προς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε προσπάθειες βελτίωσης αυτής της επικοινωνίας. Τα επόμενα χρόνια θα πρέπει όλοι να δουλέψουν για μια κοινή μεταναστευτική ε, πολιτική έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα ε, που αντιμετωπίζει ήδη η κοινωνία. Τώρα περιμένω τα σχόλιά σας, τα οποία θα ληφθούν υπόψη στον προπαρασκευαστική μας εργασία για την νέα Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, εν τέλει να πω ότι βεβαίως είμαστε πάντα στη διάθεση της Επιτροπής σας έτσι ώστε ε, να ε, γίνει σε βάθος συζήτηση εδώ στην Ολομέλεια οποτεδήποτε μας το ζητήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Ελ για την ενημέρωση. Σωστά το είπατε ότι αυτή η ενημέρωση χρειάζεται κυρίω για τους νέου συναδέλφου αλλά και για όλους γενικότερα και σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε σε όλα τα θεσμικά όργανα μπορούμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να βλέπουμε που υπάρχουν τα παραθυράκια, τα προβλήματα, οι ελλείψεις. Αυτά πρέπει να τα επισημαίνουμε και να τα διορθώνουμε στα νομοθετήματα που έχουμε θεσπίσει. Θα πρέπει αυτά τα νομοθετήματα να εφαρμοστούν. Ακόμα και με επίκληση της διαδικασίας επί παραβάση. Να κινεί τη διαδικασία αυτή η Επιτροπή για όσο κρατημήλια δεν κάνουν το καθήκον τους. Αυτές οι οδηγίες αποσκοπούν να καλύψουν την νόμιμη μετανάστευση σηκώνει ζήτηση το θέμα, οπότε όποιος συνάδελφος θέλει μπορεί να λάβει το λόγο. Κυρία Τρίκ. Thank Πρώτη Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και τον κύριο Ελ για την ε, ενημέρωση, λέει η κυρία Στρίκ. Με αυτή τη γνωμοδότηση φαίνεται ότι πρέπει να βελτιωθεί και από πλευρά εφαρμογή, αλλά και αν χρειάζεται καινούργια νομοθεσία. Και η κυρία Φοντελάιεν μας διαβεβαίωσε ότι θα μας παίρνει στα σοβαρά. Αυτό ενθαρρύνει. Και εγώ ως πανεπιστημιακός έχω εμπλακεί σε τέτοιου είδους ε, μελέτες και έχω κάποια ερωτήματα για την νέα νομοθεσία και για την εφαρμογή. Για την εφαρμογή, όπως είπατε, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκήσει τα καθηκοντά της ως ε, ε, όργανο εποπτείας και να επικαλεστεί τη δικασία επί παραβάση. Για πες να μας κύριε Έλλον, τι έχει κάνει, τι, τι παρεμβάσεις έχει κάνει για την νόμιμη μετανάστευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για καλύτερη εφαρμογή επίσης, για πέστε μας σκοπεύετε να εκδώσετε κάποιο είδου πρακτικές κατευθυντήριες για την εφαρμογή στην πράξη, ιδίω για την επανένωση των οικογενειακών. Έχει γίνει ε, το, το, το αλλά ίσως χρειάζονται περισσότερε λεπτομερείς ε, κατευθυντήριε. Επίσης, νέα νομοθετήματα. Τρία ερωτήματα για τις ε, οδηγίες για την επανένωση. Δεν έχουμε ακόμα κάποιον ορισμό του τι γίνεται με την επικουρική προστασία. Δεν τα προβλέπει η οδηγία. Και σε επόμενες οδηγίες θα πρέπει να υπάρχουν ανάλογες διατάξεις όπως και για τους πρόσφυγες. Τι θα κάνετε για αυτά, πώς θα άρετε αυτό το κενό, γιατί βλέπουμε ότι στα κράτη-μέλη είναι θέμα το οποίο έχει σημασία, ιδίω για την επανένωση οικογενειών, οικογενειών αυτή, η επικουρική προστασία. Χρειάζεται μακρόπνοη προστασία. Χρειάζεται αυτό το μέσο. Να κρυθεί να χρήζουν προστασίες ως πρόσφυγες επικουρικής προστασίας. Πέραν βέβαια των όσων λέει ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τώρα όσον αφορά την ε, μακρά διαμονή και τη σχετική διαδικασία, έχουμε τώρα αυτή την 20η επέτειο, γιατί είπαμε ότι συγκρίσουμε δικαιώματα. Πρέπει να του απονεμηθούν όπω στοχεύει αυτή η οδηγία και σε σχέση με την κινητικότητά του δικαιώματα. Και διαπιστώνεται από την οδηγία ότι υπάρχουν φραγμοί στο να απολάβουν αυτών των δικαιωμάτων. Υπάρχει αυτό το κριτήριο της εργασίας, αλλά είναι δύσκολο τελικά αυτοί που διαμένουν επί μακρόν σε κράτος μέλος να πάρουν σε άλλο για να διαμείνουν. Αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί με νέα νομοθεσία. Συμφωνείτε κύριε Ελ, συμφωνεί η Επιτροπή, συμφωνείτε μαζί μας ότι πρόκειται περί φραγμού όσον αφορά την άσκηση των σχετικών δικαιωματών, όσον αφορά την νόμη ε, μετανάστευση, βλέπουμε ότι υπάρχει πολυνομία και υπάρχουν πολλά παραθυράκια, πολλά κενά. Είναι και θέμα αγοράς εργασίας, υψηλές ε, δεξιότητες κλπ. Τι λέτε κύριε χρειάζεται κάποιο είδους ε, σφαιρική ρύθμιση για να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες. Κυρία Στρίκ, όλα αυτά σίγουρα τα έχει σημειώσει ο κύριος Σόλη. Όλα αυτά τα προβλήματα έχουν επισημανθεί και λαμβάνονται υπόψη. Κύριε Θόητο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Διευθυντή. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα που μας ανέπτυξε σήμερα το πρωί. Και συμφωνώ στην έκθεση θα πρέπει να αναδειχθεί το πόσο χρειάζεται, να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες για να μπορέσουμε να εδραιώσουμε αυτά τα προβλεπόμενα δικαιώματα και κάποιες διαδικασίες για την εφαρμογή της νομοθεσίας μας και βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας από τα κρατη Θα πρέπει να παραδειχτούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Θετικά. Ακόμα όμως δεν έχουμε όλα τα μέτρα, όλες τις διαδικασίες και επίσης τις κυρώσεις για μη τήρηση των προβλεπωμένων. Τώρα εγκατακλείδη μια γενικότερη σκέψη μου γιατί στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ε, μα ήρθε να ζητήσουμε ε, η Κομισιόν και το Συμβουλίο να άρουν κάποιο είδους ε, ε, παραθυράκι που υπάρχει. Λέτε ότι γίνεται όσον αφορά την αγορά εργασία και του υπηκόου των χώρων. Η ρύθμιση θα πρέπει να λάβει υπόψη το εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών όσον αφορά το πώ οι υπηκοτοί των χωρών γίνονται δεκτοί, αλλά και από την άλλη μεριά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ό,τι έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε όσον αφορά την ε, μεταναστευτική πολιτική των τρίτων χωρών. Ευχαριστώ, λέει ο Ζήπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να είμαι ειλικρινής, ως πεπειραμένο μέσα αυτής της Επιτροπής και έχοντας υπόψη ότι δεν έχει την αποκλειστική ευθύνη η Κομισιόν, δεν, παρόλα αυτά ε, δεν έχω εντυπωσιαστεί από αυτήν την παρουσίαση και έχω ερωτήσεις. Σε πρώτη, μιλάμε για την εφαρμογή οδηγιών που είναι από το 2003 και το 2011. Υπάρχει έστω και μια χώρα που πλήρως να εφαρμόζει αυτές τις οδηγίες. Δεύτερον, μιλούμε για οδηγίες. Άρα, ο τρόπος εφαρμογής μπορεί να είναι ε, πολύ διαφορετικό σαν κράτο μέλος και αυτό ισχύει και στην πράξη. Βλέπετε λοιπόν κάποια ε, βήματα να γίνονται προς την εναρμόνιση των κανόνων σε οποιαδήποτε χώρα ή οι κανόνες εξακολουθούν να είναι εντελώ διαφορετικοί στα 28 κράτη-μέλη. Αν δει κανείς ε, τις διάφορες κατηγορίες εργαζομένων και τους κανόνες, γιατί νομίζω αυτό το ήθελε το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη. Πόσο δύσκολο θα είναι για επικός τρίτων χωρών να καταλάβουν ποιοι κανόνες τους αφορούν και σχετίζονται με τις δικές τους επιθυμίες και πόσο πολύπλοκο είναι να καταλάβει κανείς τι πρέπει να κάνει για να ε, θεωρηθεί νόμιμος μετανάστης και να αναζητήσει ε, εργασία σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται κάποια συζήτηση, υπάρχει κάποια πρόθεση σε επίπεδο ε, επιτροπής για να υπάρξει κάποια εναρμόνιση στο τέφα την νόμιμη μετανάστες. Και ο τρίτος τομέας είναι η επανένωση των οικογενειών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βασίζεται μόνο στο κράτος δικαίου επιμένουμε ότι είμαστε και ήπειρος η οποία δράζεται σε θεμελιώδη δικαιώματα και η επανένωση των οικογενειών φυσικά και είναι ένα πολύ σημαντικό δικαίωμα. Είναι και πολύ σημαντικό και στο πίσω τη χριστιανικής μας παράδοσης η οικογενειακή επανένωση όμως δεν είναι κάτι εύκολο. Και σε ό,τι αφορά την νόμιμη μετανάστες και σε ό,τι αφορά το άσυλο. Έχουμε ένα επιδείξουμε κάποια επιτυχία σε αυτό το μέτωπο <coughs> και αν έχει επιτευχθεί πρόοδος πού. Πάντως δεν νομίζω ότι υπάρχει και πολύ εναρμόνιση και στα λέω, σας τα λέω ανοιχτά. Κάποιοι λένε ότι ίσως χρειάζονται άσυλο και φτάνουν εδώ όμως όχι γιατί πραγματικά θέλουν να ζητήσουν άσυλο, αλλά γιατί δεν έχουν προοπτικές στη χώρα τους και ψάχνουν δουλειά. Γιατί όμως επιλέγουν αυτό τον επικίνδυνο και ενδεχομένως μοιραίο για τη ζωή τους ε, τρόπο. Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι. Ίσως η περισσότερη εναρμόνιση θα βοηθούσε καλύτερα από το να επιμένουμε σε εθνικά στοιχεία, εθνικά μέτρα. Από το 2003 και ε, μέχρι τώρα τι έχει γίνει. Έχουμε 28 για να μην πω εκατοντάδες διαφορετικά ε, εργαλεία, συστήματα ή υπάρχει κάποια εναρμόνιση. Πρόεδρος, κύριε Έλλη βλέπετε ότι διευρύνθηκε πλέον ε, το θέμα και δεν υπάρχει μόνο η διάθεση αυτοκριτικής, αλλά όλοι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. ερωτήσει. Βλέπω και τον κύριο Βάιμερ που θέλει να πάρει το λόγο. Thank you, uh, Mr. Chairman. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, προς την κυρία Ελ. Καλό είναι που κάνετε αυτές τις εκτιμήσεις, αλλά καλύτερα θα ήταν να ελέγξετε περισσότερο ποιες είναι οι συνέπειες και πτώση του να υπάρχει λιγότερη ρύθμιση στον τομέα αυτό. Καλό καλοδεχούμενο αυτό που είπατε για την οδηγία περί πανένωσης οικογενειών. Δηλαδή, ότι οι περισσότεροι από που παίρνουν άδειε παραμονή είναι μέλη οικογενειών ε, μεταναστών. Στη Σουηδία, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, αυτό σημαίνει ότι εμείς σε αιτήσια βάση λαμβάνουμε ή χορηγούμε πάνω από 100.000 άδειε παραμονής. Παρά το γεγονός που το... το ότι η κυβέρνηση ε... έδωσε άλλες υποσχέσεις, ότι θα μειωθεί δηλαδή ο Τι δυνατότητες υπάρχουν. Έχετε τη βούληση να περάσετε από αυτό το σύστημα σε ένα σύστημα gastarbeiter κατά κάποιο τρόπο που να μην είναι τόσο εύκολο να φέρνει κανείς όλη την οικογένεια και το σόι του μαζί. Έχετε ζητήσει το λόγο εσείς, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστώ τον κύριο Ιούλη. Θα είμαι πολύ σύντομο στο ερώτημα που θέλω να θέσω. Διάβασα και τα έγγραφα. Και είναι και κατατοπιστικά για μένα ως νέο βουλευτή. Δεν έχω την εμπειρία της κυρίας Ζίπελ, αλλά ε, αν κατάλαβα καλά αυτά που είπε, μίλησε για το σήμερα. Εγώ έχω μια συγκεκριμένη πρόταση που έχει να κάνει με την επιβολή της εφαρμογής αυτής της νομοθεσία σε επίπεδο κρατών μελών. Έχετε προτάσεις για την ενίσχυση επιβολής νομοθεσίας για το μέλλον. Γιατί είναι κάτι σημαντικό. Στο οποίο το λέω κατά Ευχαριστώ. Ο κ. Σασμάνη από την Άλτη ήταν αυτός που ακούσαμε, δεν υπάρχει κάποιο άλλο. οπότε θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ελ. Περιμένουν οι συνάδελφοι απαντήσεις, κύριε Ελ, στα συγκεκριμένα ερωτήματα που σα έθεσαν. Έχετε το λόγο. Uh, um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλές παρατηρήσεις, ε, πολλές ερωτήσεις. Χαίρομαι γι' αυτό. Το είπα και στην παρουσίασή μου ότι τώρα προβληματιζόμαστε, σκεφτόμαστε για το πώς θα ε, παρουσιάσουμε το όλο θέμα υπόψη της νέα ε, Επιτροπής και σε αυτά τα πλαίσια βέβαια θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις σας. Για την κυρία Στρίκ, πολλές ερωτήσεις για την υλοποίηση και τις ε, ελλείψεις ε, ε, όσον αφορά την υλοποίηση. Εδώ μιλάμε για οδηγίες που θα πρέπει να μεταφερθούν στο δίκαιο, να εφαρμοστούν από τις χώρες. Υπάρχει ακόμα και αυτόματη διαδικασία για άμεση έναρξη διαδικασίας επί παραβάση εάν δεν ε, υλοποιηθεί σωστά, εάν ε, δεν έχει ειδοποιήσει την Κομισιόν ότι ε, πλέον εφαρμόζει την οδηγία κλπ. Επίσης αναφέρατε ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν ε, γνώση ε, και, δεν, και χρειάζονται κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Δεν είναι γεγονός ότι θέλουμε να ενισχύσουμε τις ε, κατευθυντήριες γραμμές και να τις κυκλοφορήσουμε περισσότερο. Επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορώ να, πω, ε, σε, να μπω σε πολλές διαπραγματεύσεις, συγγνώμη σε πολλές λεπτομέρειες, ε, γιατί το θέμα ε, των διαδικασιών επί παραβάση για τον τομέα αυτό βρίσκονται τώρα στο τραπέζι των συζητήσεων. Επίσης αναφερθήκατε στην, ε, ε, στην προστασία των ε, τον άσυλο και στην επικουρική προστασία. Να σας πω ότι ο έλεγχος καταλληλότητας έχει καταλήξει ότι υπάρχει κάποια διαφορά όσον αφορά τους ε, δικαιούχους ε, άδεια παραμονής ε, και τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας. Θα το δει το θέμα αυτό η επόμενη Επιτροπή και οι συνομοθέτες. Πάντως αυτό το οποίο αναφέρατε όντως έχει καταδειχθεί και στο fitness check όσον αφορά την οδηγία για την άδεια ε, παραμονής ε, για τους διαμένοντες για μεγάλη διάρκεια. Κάνατε διάφορες προτάσεις, ε, καταγράφονται αυτές, δεν χρειάζεται να μπω εδώ σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο κύριος Θοίδο, είπατε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι θετικές εξελίξεις που έχουν επιτευχθεί. Πρέπει να σας πω ότι στην έκθεση εμείς έχουμε ε, αναφέρει χαρακτηριστικά και για το θέμα αυτό αναφερόμαστε ε, και στις ελλείψεις όσον αφορά τα εργασιακά και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, τους στόχους ε, της πολιτικής νόμιμης μετανάστευσης. Και να πω κύριε Πρόεδρε ότι η πολιτική νόμιμης μετανάστευσης έχει τρεις διαφορετικούς πυλώνες. Για κάθε πυλώνα θα πρέπει να σκεφτούμε τα επόμενα χρόνια πώς θα βελτιωθεί. Ο πρώτος πυλώνας είναι η ενωτική ε, πλευρά, ε, σχετίζεται με την ε, τον επαναπατρισμό ή το resettlement και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτός ο πυλώνας είναι σωστός και είναι ο ανθρωπιστικός πυλώνας. Δεύτερος πυλώνας είναι ε, αυτός που σχετίζεται με την αγορά εργασίας. Είναι οι μπλε κάρτες και εδώ πρέπει να δούμε πόσο και πού θα προχωρήσουμε είναι ανοιχτά πολιτικά ζητήματα αυτά. Τρίτος πυλώνας που δεν πρέπει να λησμονούμε είναι το εξής. Εάν δεν έχουμε συλλογική, συνολική μάλλον ευρωπαϊκή πολιτική, παρόλα δεν δεν μπορούμε να προσφέρουμε σχεδόν τίποτα στις τρίτες χώρες στη διαπραγμάτευση όσον αφορά τις επιστροφές ε, ε, και τις επαναπροωθήσεις. Ε, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την παράτυπη μετανάστευση, αλλά ταυτόχρονα πρέπει κάτι να προσθέσουμε, να προσφέρουμε. Θα πρέπει να δώσουμε τα νόμιμα, της δυνατότητες συγγνώμη, για νόμιμη μετανάστευση. Αυτά σε σχέση με τον κύριο Θοήδο. Η κυρία Ζίβελ αναφέρατε πολλά σημεία τα οποία είναι πολιτικά ε, και επομένως ε, πρέπει να σας ε, παραπέμψω στην επόμενη πολιτική στην επόμενη Επιτροπή, γιατί αυτά θα πρέπει να συζητηθούν από πολιτική άποψη. Στην έκθεση εμείς λέμε ότι υπάρχει πραγματικά ε, πρόβλημα ε, εφαρμογής, ε, υλοποίησης των προηγούμενων παλαιών οδηγιών. Επομένως δεν μπορείτε να μου λέτε ότι τα βλέπουμε όλα ροζ και χαριτωμένα καθόλου. Αναφέρουμε όλα τα προβλήματα όσον αφορά την αυξημένη, ε, τον αυξημένο εναρμονισμό, αυξημένη εναρμονισμό των κανόνων. Θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πολιτική κατάσταση και ποια θα είναι η πολιτική θέση και της επόμενης Κομισιόν. Και αυτό απαντά και την τελευταία παρέμβαση που αναφέρθηκε στην αδυναμία ε, διαφορετικής νομοθεσίας. Ε, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι απήντησα στις κύριες ερωτήσεις, τουλάχιστον απήντησα σε αυτές τις οποίες είμαι σε θέση να απαντήσω τώρα. Πάντως, εάν θέλετε ως Επιτροπή να έχετε πιο τεχνική συζήτηση και όσον αφορά τα αποτελέσματα αυτού του fitness check, του ελέγχου καταλληλότητας, βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Όλε, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, ναι, θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να συζητήσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά στοιχεία ε, της, και αυτές τις πτυχές της μεταναστευτικής πολιτικής. Ε, πολλές φορές αναφέρεται ότι ναι υπάρχουν κάποια νόμιμα εργαλεία στη διάθεση αυτών που θέλουν να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη αλλά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για όποιον θέλει να φτάσει στην Ευρώπη. και επομένως πρέπει να δούμε στο σύνολό της ε, την ε, πολιτική μετανάστευση και φυσικά είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει την ε, Επιτροπή μας εδώ, την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ολοκληρώσαμε τα σημεία που είχαμε στην ημερήσια διάταξη. Τρεις η ώρα σας περιμένουμε εδώ. Θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον Julian King, Επίτροπο Αρμόδιο για την Ένωση ασφάλειας, θα μας μιλήσει για τη στρατηγική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα χρόνια. Όμως, να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε συνεδρίαση των συντονιστών σε λίγα λεπτά, αλλά όχι εδώ, όχι εδώ, θα αλλάξει η αίθουσα. Στην ε, ε, Αλτιέρο Σπινέλη, ή 2. Ή 2 λοιπόν και θα ξεκινήσουμε στις 11.30 και θα διαρκέσει η συνεδρία των συντονιστών μέχρι τις 12.30. Θα ξαναρχίσουμε ως Επιτροπή της Εργασίας μας στις 3 το απόγευμα, παρακαλώ. Χαίρετε.